συγκεκριμένες ε, περιπτώσεις που δεν ε, αναφέρονται πολύ συχνά μιλώντας για φυλακές ε, αλλά όχι για τους τρομοκράτες θα ήθελα να θυμίσω τις συνθήκες τις απάνθρωπες των φυλακών στην Ρουάντα και στη Λιβύη όπου η θανατική ποινή είναι μια πρακτική στην κράτηση ανθρώπων που δεν έχουν κανένα ε, δεν έχουν διαπράξει κανένα έγκλημα. Να θυμίσω επίση την υπόθεση των Σαχαραουί, η οποία δεν έχει ακόμα επιληθεί εδώ και τόσα χρόνια και να θυμίσω επίση πω υπάρχουν ε, δικαιώματα για του πρόσφυγε λόγω κλιματικών αλλαγών που διώκονται από τη χώρα του, οθούνται μάλλον εκτό τη χώρα του, λόγω των δραματικών κλιματικών αλλαγών. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη γιατί ακριβώ αποτελούν την βάση και τη δική μα συμβίωση. Ευχαριστώ. Ο κύριος για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για την 60η επέτειο των ΟΗΕ το 2005 δημιουργήθηκαν νέε δομέ. καταρχάς το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και η Επιτροπή ε, Ειρνευτικών Δυνάμεων. Η Επιτροπή αυτή ε, συνέχισε το έργο τη ε, επαρκώ. Το ίδιο δεν μπορούμε να πούμε ότι το Συμβούλιο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και αυτό εκφράζουμε στο ψήφισμα, ότι χρειαζόμαστε κατεπηγόντω μία μεταρρύθμιση για να μην είναι τόσο μονόπλευρο το έργο του Συμβουλίου Ανθρώπινων Δικαιωμάτων. Αυτό λοιπόν δεν έχει θυχτεί επαρκώς και χαίρομαι και λυπάμαι που το τονίζει, δεν το τονίζει αυτό α, επαρκώς το Συμβούλιο. Λέει ο συνάδελφος Χάουαρτ ότι θα πρέπει, αν εκλεγεί το Ιράν, θα είναι αυτό ε, θα αντιφόρο χτύπημα για το Συμβούλιο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων. Θα πρέπει να μας πει τι σημαίνει αυτό. Γιατί νομίζω ότι αν συνεχίσουμε κατά αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να εξετάσουμε πάρα πολύ σημαντικά με το θέμα της Επιτροπής των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στα Ηνωμένα Έθνη που έχουν ε, διεθνή εκπροσώπηση και υψηλότερο ε, κονδύλιο. Το ξέρετε και το ξέρουμε ότι το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι μια μεγάλη δύναμη. Ε, ξέρουμε ότι από την άλλη πλευρά υπάρχει το θέμα, το πρόβλημα μάλλον ε, της ε, Συνόδου των Ισλαμικών χωρών. που ε, Είναι ένα σώμα το οποίο θέλει να βάλει κατά του Ισραήλ και το Ιράν είναι αυτό που το υποστηρίζει. Είναι είναι απίστευτο που παίρνουμε στα σοβαρά αυτό το Συμβούλιο. Αν πραγματικά στα σοβαρά θέλουμε να μιλήσουμε για ανθρώπινα δικαιώματα ως Κοινοβούλιο, θα πρέπει να αντιτεθούμε στην παραβίαση, την κατάφορη παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων από πλευρά των χωρών που βρίσκονται σε αυτό το Συμβούλιο, Αραβία, ε, Πακιστάν, Ινδονησία, Αίγυπτος, παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και βρίσκονται στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Μα τώρα θέλει να μπει και το Ιράν. Ε, τι λείπει, η Βόρειος Κορέα θα είναι όλοι μαζί με τα παρέα. Πρόεδρε, γιατί ο κόμμα μας είναι ξεκάθαρο. Το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι ένα πολύ τρομακτικό όργανο που δεν μπορούμε να το παίρνουμε στα σοβαρά. Θα πρέπει πραγματικά να κρατήσουμε τις αποστάσεις μας από αυτό το Συμβούλιο και να μην ε, αντιφάσκουμε με την δική μας πολιτική για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα αρχίσω υπενθυμίζοντας ότι όταν ιδρύχεται το ενιαίο για τα ανθρώπινα δικαιώματα μέσα στο Ηνωμένη Έθνη, το Συμβούλιο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ήταν η πραγματοποίηση μιας ελπίδας για την καλύτερη προστασία των βασικών δικαιωμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο. Ε, η μέθοδος ε, περιοδικών εξετάσεων σε όλο τον κόσμο ήταν μια καινοτομία που θα είχε σαν στόχο να ανταποκριθεί στην συνεχή πολιτικοποίηση της καταπολέμησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και έτσι για να μπορέσει το Συμβούλιο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να πληρώσει την εντολή του, βλέπουμε ότι οι παλιοί δαίμονες εξακολουθούν να δρούν. Ο μηχανισμός παγκοσμίου ελέγχου περιοδικού ελέγχου δεν αρκεί για να προστατευτούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, γιατί αν το Συμβούλιο δεν αντιδράσει αρκετά γλίγορα, όπω έγινε παραδείγματο χάρη στην Γουινέα, αυτό έχει επιπτώσεις σημαντικότατες. Όποιος δεν σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα βρίσκεται ατιμόρυτος. Γι' αυτό πρέπει να αντιδρούμε αυστηρά και γλίγορα για την καταπάτηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Θα πρέπει λοιπόν η Ένωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προωθήσει τους μηχανισμούς ανταποκρίσης της κρίσης όπως το Αφγανιστάν, στη Γενέα, στην Ιράν, στην Ιεμένη και στο Ιράκ. Έχει όφελο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να είναι το πιο ισχυρό και το πιο αποτελεσματικό δυνατόν, γιατί χρειάζομαι νομίζω έναν δραστήριο εταίρο στον τομέα αυτό. Ευχαριστώ. Αγαπητέ Επίτροπε, Αγαπητοί συνάδελφοι, εγώ θα, ήθελα να σας μιλήσω για κάτι που αποτελεί διαρκή ανησυχία όσον αφορά την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κυρίως ε, μετά από την κατάσταση που δημιουργήθηκε ε, μετά από τον ε, σύγκρουση στη ε, περασμένο χειμώνα και τα δύο μέρη ε, προκάλεσαν ε, προβλήματα για τον ε, πληθυσμό, τον άμαχο πληθυσμό στο Ισραήλ και στην Παλαιστίνη. Είναι δύσκολο να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Οι επιθέσεις της ΑΜΑΣ δεν, μπορεί, δεν έκαναν τίποτα άλλο παρά να τρομακροτήσουν τους άμαχους του Παλαιστίνης και του Ισραήλ. Γνωρίζουμε τα δύο μέρη και πιστεύω πως δεν θα πρέπει να προσπαθήσουμε να ενοχοποιήσουμε τον έναν, τη μία μονοπλευρά. Οι πρακτικές και ανθρωπιστικές συνέπειες όλων αποτελούν ε, ένα ε, μια έκκληση ε, για να προσπαθήσουμε να λύσουμε παγκόσμια αυτή την, αυτή την σύγκρουση και να προωθήσουμε τον διάλογο για την ειρήνη. Είναι ένας τομέας όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την απαραίτητη την αξιοπιστία για να ενεργήσει και να ενεργήσει με πιο σταθερό τρόπο. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε κύριε Υπουργέ. Μία από τις ε, κοινοβουλευτικές προτεραιότητες είναι να αντιμετωπίζονται ανισχυτικές καταστάσεις όπως δραστηριότητες ε, που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν πολιτικοποιηθεί πλήρω. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική τα μέλη της Αντιπροσωπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ε, ζητήσουν να πληρωθούν τα κριτήρια για να μπορέσουν να γίνουν μέλη του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών. Γιατί έτσι μπορούν να αντιμετωπίσουν την χρήση ε, αποφάσεων για μη δράση, για αδράνεια, σε περιπτώσει καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα ήθελα να αναφερθώ επίση σε δύο κοινοβουλευτικέ προτεραιότητε. Καταρχήν, Λευκορωσία. Εν αντιθέσει από τι ε, προσδοκίε, η κατάσταση για τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν βελτιώθηκε. Επιδεινώθηκε μάλιστα. Θα ήθελα να τονίσω το μήνυμα του κ. Μανικέβιτς σήμερα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τώρα τη δυνατότητα να ασκήσει πίεση στο καθεστώς Λεκοσέγκο για να μπορέσει να προωθήσει βελτιώσεις και αλλαγές σαν προϋπόθεση για την χορήγηση οικονομικής βοήθειας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ την ε, δήλωση της περισμένης εβδομάδας 18 ε, ατόμων που δρούν υπέρ των ανθρώπινων δικαιωμάτων στην ε, Ρωσία, μεταξύ αυτών και ο κάτοχος του Συμβουλίου του βραβείου συγγνώμη Ζαχάροφ, είναι πραγματικά πάρα πολύ κακό για, τις, για την εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επενούν ανθρώπους όπως τον κύριο Καβάλιοφ που του δώσαν το βραβείο Ζαχάροφ και από την άλλη μεριά να υποστηρίζουν τον κύριο Πουτίν στην πολιτική που ασκεί. Ευχαριστώ. Του ε, η κυρία Μπασέσκου για ένα λεπτό. Θα ήθελα να αναφερθώ στην περίπτωση του Γιλιά Σαλίτ, στρατιώτη Ισραηλινού, που εξαφανίστηκε τον Ιούλιο του 2006. Ένα στρατιώτης 19 ετών μόλι. Την περασμένη εβδομάδα ήμουν τμήμα τη επίσημη αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Ισραήλ και συναντήσουμε τον ε, πατέρα του κ. Σαλίτ, τον κ. Ραμασολέτ. Παρόλα τα άρθρα 13, 23 και 126 της Σύμβασης της Γενέβης όσον αφορά τα δικαιώματα των ε, των πολέμων ο Γιλάτ που έχει και τη γαλλική υπηκότητα δεν έχει το δικαίωμα να δεχθεί η... τα από την οικογένειά του ούτε από τον Ερυθρό Σταυρό, οι οποίοι δεν γνωρίζουν καν πού βρίσκεται. Θα ήθελα να διευκρινίσω ότι το άρθρο 77 της έκθεσης Κόλστον που επικρίνει το Ισραήλ αναφέρει ότι ο Γιλασαίτ θα πρέπει να ωφεληθεί από τα δικαιώματα της συνθήκης της Γενέβης και ζητά από την, Γενέβη, από την να δεχθεί τα δικαιώματα αυτά. Az EU az ki kell fejezze abéli meggyőződését, θα πρέπει σαφώ να πούμε στο ψήφισμά μας, ε, κατά την άποψή μου, ότι γίνονται παραβιάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στι αναπτυσσόμενες χώρε αλλά το ίδιο συμβαίνει και στις ανεπτυγμένες. Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και η δήλωσή του του 1992, 18 Δεκεμβρίου, δηλώνει, ορίζει μάλλον τα δικαιώματα των εθνικών, εθνοτικών, θρησκευτικών, ε, άλλων μειονοτήτων και αυτό ισχύει τόσο για αναπτυσσόμενες χώρες όσο και για τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, η δεύτερη παράγραφος δηλώνει σαφώς ότι Εθνικές μειονότητες ε, δικαιούνται να χρησιμοποιούνται τη μητρική τους γλώσσα στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα χωρίς να πέφτουν θύματα οποιασδήποτε παρέμβασης ή διάκρισης. Ε, και αυτή η διάταξη θα πρέπει να τηρείται και από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αξιόπιστη εάν βρει λύση για το πρόβλημα αυτό και εισάγει μέτρα τα οποία να ε, τηρούν υποδηματικά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Τα επόμενα δύο χρόνια, κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, είναι κρίσιμα για την αποκριστάλλωση του ρόλου του ΟΗΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, γιατί όπω είναι γνωστό, το 2011 θα δει το φω τη δημοσιότητα η διακυβερνητική επισκόπηση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Υπάρχει κίνδυνο σε αυτό το διάστημα χώρε οι οποίε αναφέρθηκαν και από του συναδέλφου και οι οποίε δεν αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στον τομέα αυτό να προσπαθήσουν να περιορίσουν το ρόλο του ΟΗΕ σε όσα ήδη αναφέρθηκαν προσθέτω τα εξή πρώτον εφόσον η ευρωπαϊκή ένωση είναι και επιθυμεί να συνεχίσει να είναι ένα από του σημαντικότερου παράγοντε όσον αφορά στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μια από τι προτεραιότητέ μα πρέπει να είναι να μιλάμε διεθνώ με μια φωνή και να αποφεύγουμε όσο μπορούμε τι παραφωνίε. δεύτερον θα πρέπει να ενισχύουμε και τη συνεργασία μα με τι ηνωμένε πολιτείε τη αμερική στον τομέα τη προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. και τρίτον και τελευταίο το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο πρέπει και μπορεί να παρακολουθεί προσεκτικά τι ειδικέ διαδικασίε που θα ακολουθήσουν όσον αφορά την καθολική περιοδική εξέταση του συμβουλίου ώστε να υπάρξει πραγματική ουσιαστική συμβολή από την πλευρά μα στην προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλα τα κράτη μέλη των ηνωμένων εθνών. ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Η κυρία Νελτζέλτσοβα, για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Γκαριό, κύριε Λαμπρό θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σα στο ψήφισμα, σημείο 13, όσον αφορά την υποψηφιότητα για το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Τη ε, περασμένο καλοκαίρι εξετάστηκε η τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν. Το καθεστώ του Ιράν επιβεβαιώσε ότι εξασφαλίζεται ο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα αυτή. Θα ήθελα αυτή τη στιγμή να τονίσω όμω κάτι διαφορετικό. Η χθε η κυρία Μαρία Μιρατζεβί μα παρουσίασε τι. Ε, ε, και βασανιστήρια σε γυναίκες στο Ιράν που είναι κατά του καθεστώτος. Είναι χαρακτηριστική αυτή η καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επίσης άλλες ματριές ακούσαμε τον Γενάρη. Δεν μπορούμε να δεχθούμε σήμερα το Ιράν να γίνει μέλος του Συμβουλίου της, των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στον ΝΟΕ. Γιατί αλλιώς πώς θα σεβόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα πρέπει να μιλήσουμε με μία φωνή η Ευρωπαϊκή Ένωση. όπω η κυρία Σόλα θα πρέπει να μην ληφθεί καν υπόψη η υποψηφιότητα του Ιράν εδώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόεδρε, Αυτές οι παραβιάσεις των ανθρωπινών δικαιωμάτων αφορούν μια σειρά χωρών εδώ. Και είναι πάρα πολύ σοβαρές. Εγώ θεωρώ ότι ο ΙΕ εδώ και καιρό έχει κρίνει επ' αυτόν. Επομένως, θα πρέπει να λάβουμε δράση κατά αυτών των παραβιάσεων θα πρέπει επομένω να κατονομαστούν οι παραβάτες. Θα πρέπει ξεκάθαρα να στείλουμε το μήνυμα ότι είναι απαράδεκτες αυτές οι συστηματικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει προς αυτή την κατεύθυνση που έχει αποφασιστεί με τα ψηφίσματα. Είναι ο Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οι χώρε στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει πρώτα-πρώτα να κοιτάξουν τα του οίκου του, το περιβόλι του, πριν κατηγορήσουν του άλλου γιατί. Πάρα πολλά τέτοια κράτη διώκουν και φυλακίζουν. Κάποιους κατά της ελευθερίας του λόγου. Επίσης κατάσχονται βιβλία, απαγορεύουν όπως το Βέλγιο κάποια πολιτικά κόμματα και στο Βέλγιο και στη Γερμανία. Και πολλές φορές αυτό γίνεται συγκαλυμμένο όπως γίνεται στη χώρα μου. Το δικό μας κόμμα απαγορεύτηκε με δικαστική απόφαση και απαγορεύτηκε να γράφουμε μέλη επαορίστο. Λέγονται δημοκράτες, αλλά θα πρέπει να σεβαστούν και το δικαίωμα του λόγου, του συναθρίζεστε, αλλά και του εκλέγει και εκλέγει. Ευχαριστώ πολύ και τώρα για να κλείσει η συζήτηση εξ ονόματος του Συμβουλίου ο κύριος Λόπες Καρίδο. Gracias, señor presidente. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ε, ευχαριστώ όλους όσοι έλαβαν τον λόγο για το θέμα το οποίο τώρα συζητούμε που είναι σημαντικό. Είναι ένα από τα βασικά στοιχεία όπως προείπα για την ευρωπαϊκή πολιτική για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εμείς θέλουμε να εμπλακείτε όλοι, να μας βοηθήσετε στην υπόθεση αυτή. Θα πρέπει η γραμμή μας πλεύσης να συνεχιστεί γιατί ανέκαθεν θέλαμε να υπάρξει ένα τέτοιο Συμβούλιο Ανθρωπινών Δικαιωμάτων το οποίο να αντικαταστήσει την Επιτροπή Ανθρωπινών Δικαιωμάτων. Κατά τη γνώμη μας είναι ένας φορέας, ένα όργανο το οποίο μπορεί επαρκώς να χειριστεί τέτοιες περιπτώσεις παραβίασης των σε όλο τον κόσμο. Περιπτώσεις που απαιτούν ανάληψη δράσης και αντίστοιχη αντίδραση και τοποθέτηση και του ΟΗΕ. Γι' αυτό σας λέμε ότι η Προεδρία του Συμβουλίου της Ένωσης ανέκαθεν και συστηματικά το στις συναντήσεις του Συμβουλίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό θα συνεχίσουμε και να το πράττουμε. Στην επόμενη σύνοδο του Συμβουλίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα είμαστε εκεί ως ε, Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρούμε ότι κάτι τέτοιο συμβαδίζει με τόσο έχουμε δηλώσει, με τις τοποθετήσεις όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης, σας βεβαιώνουμε ότι θέλουμε να συνεχίσει να υπάρχει ένας τέτοιος φορέας και έτσι να μπορέσουμε να εξαντλήσουμε τις δυνατότητες που παρέχονται. Προς το παρόν, σε μερικές περιπτώσεις ε, τις εκμεταλλεύουμε, σε μερικές περιπτώσεις όχι. Ε, έχουμε βέβαια και τις σχετικές ψηφοφορίες. Δεν πετυχαίνουμε πάντα το σκοπούμενο. Σε κάποιες περιπτώσεις τα πράγματα πάνε καλά, όπως ας πούμε για την Σομαλία αλλά σε άλλες περιπτώσεις δεν πετυχαίνουν αυτό το οποίο θέλουμε όμως θεωρούμε ότι οι ευτυχείς καταλήξεις των διαδημάτων μας εκεί είναι περισσότερες από τις αρνητικές αναφέρθηκαν διάφορες περιπτώσεις χωρών και στη συνέχεια βέβαια θα συζητήσουμε και για κάποιες άλλες χώρες που προβλήματα Ήδη συζητήσαμε για το Ιράν και για την σχετική του υποψηφιότητα. Όπως ξέρετε, επανειλημμένα εμείς έχουμε κάνει σχετικές δηλώσεις. Τρεις φορές μόλις φέτος. Τοποθετήθηκε σχετικά η ψηλή εκπρόσωπος, η Καθλίν, Καθλίν Άστον. Δήλωσε σχετικά με το Ιράν παραβίαση των ποινών δικαιωμάτων, δήλωσε πόσο προβληματίζεται, πόσο ανησυχεί για αυτή την περίπτωση, ε, κατεδίκασε κάποιες εκτελέσεις που έγιναν στο Ιράν. Οφείλουμε να σα πούμε ότι όσον αφορά αυτή την υποψηφιότητα είναι θέμα το οποίο είναι ακόμα θέμα εθνικής αρμοδιότητας. Το ποιο λέει δηλαδή, θα μπει στο Συμβουλίο Δικαιωμάτων. Η κατάσταση που επικρατεί στη χώρα εκείνη, οι παραβιάσεις που γίνονται και άρα το πόσο αυτά θα επηρεάσουν την υποψηφιότητα και αποδοχή της χώρας αυτής στο Συμβούλιο, αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το χειριστούμε με προσοχή για να μην καταλήξουμε σε κάποια υπερβολικά και ακραία αποτελέσματα που θα είναι αντίθετα των σκοπουμένων. Επομένω και εμεί θα πρέπει να σεβαστούμε αυτή την, την κατάσταση των πραγμάτων και να είμαστε όσο γίνεται πιο συντονισμένοι, να παρακολουθούμε τη συγκυρία, πώ κυλίζονται τα πράγματα και να είμαστε, όπω προείπα, προσεκτικοί. Τέλο, Πρόεδρε. Θεωρούμε ότι πρόκειται για ένα βήμα όπου μπορούμε να προβάλλουμε τι θέσει τη Ένωση. είναι ό,τι πιο δόκιμο υπάρχει και επομένω εμείς Θέλουμε να μην υπάρχει κανένα είδου πίσω γύρισμα όσον αφορά την πρόοδο της κατάστασης των δικαιωμάτων σε παγκόσμια κλίμακα, γιατί είναι μια κατάκτηση για όλη την ανθρωπότητα. Είναι μια παγκόσμια αξία. Είναι κάτι που θα πρέπει κανεί να το υπερασπίζει πέρα από σύνορα, παραδόσεις, ε, διαφορετικότητε. γιατί ακριβώ είναι κάτι το πολύ πιο σπουδαίο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους βουλευτές για τις συστάσεις που μας μεταβίβασαν και που είμαστε σίγουροι ότι θα τις μεταδώσουμε στην το εκπρόσωπο. Θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια συγκεκριμένα σχόλια και ερωτήσεις. Καταρχήν για την υποψηφιότητα του Ιράν. Συμφωνώ με τις απόψεις της Ισπανικής Προεδρίας. Δεν μπορώ να τονίσω ότι κάθε εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου πρέπει να παρουσιάσει στην πράξη έντονη δέσμευση για την προστασία και πρόθεση των ανθρωπινών δικαιωμάτων. Θα ήθελα να πω ότι καταδικάζουμε τη συνεχή φυλάκιση πάνω από 200, 200 αντιφρονούντων στην Κούβα. Θα μπορούσαμε να δώσουμε και άλλα παραδείγματα για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Κομισιόν καλεί την Κούβα να αλλάξει την πολιτική της, να τηρήσει υποχρεώσεις της και το διεθνές δίκαιο θα συνεχίσουμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον διάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Κούβα και με τις εκεί αρχές και θα χρησιμοποιήσουμε το διάλογο αυτό σαν ένα μέσο για να προωθήσουμε το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όσον αφορά τις ε, προσκλήσεις να μιλάει με μία φωνή η Ευρωπαϊκή Ένωση για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η Κομισιόν προφανώς το υποστηρίζει απόλυτα. Και για το θέμα για την Γάζα θα πρέπει να το αναφέρουμε στο επόμενο σημείο στην έκθεση Goldstone. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Thank you very much. Έλαβα έξι προτάσεις ψηφίσματος προς περάτωση αυτής της συζήτησης, η οποία και έληξε. Dear colleagues, as an indication of true European solidarity, not to mention humanitarian greatness towards your President, who is suffering from a terrible cold, if anyone has aspirin, you have my permission to come up here in the podium and give it to me. And I would be... Θα είμαι πολύ αυστηρός και μάλλον θα είμαι ευγνώμων σε εσάς αν κρατήσετε το χρόνο σας. Περνάμε, θα περάσουμε στο επόμενο θέμα του Συμβουλίου και της Επιτροπής για την εφαρμογή των συνστάσεων της εκθέσεως Goldstone σχετικά με το Ισραήλ και την Παλαιστίνη. Τον λόγο εξ του Συμβουλίου έχει ο κύριος Λόπες Γκαρίντο. Ευχαριστώ.